Έχουμε τη συζήτηση για τις εκτελέσεις ε, στην Αίγυπτο. Θα ξεκινήσουμε με τους συντάκτες των ψηφισμάτων. Ε, πρώτη κυρία Αντρικιένη για ένα λεπτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η Αίγυπτος έχει ε, αντιμετωπίσει δύσκολες προκλήσεις μετά την επανάσταση του 11. Η διεθνή κοινότητα στηρίζει τη χώρα στις πολιτικές οικονομικές προκλήσεις και προκλήσεις ασφαλείας. Έχουμε όμως ε, τρομοκρατικές επιθέσεις όπως στη Χερσόνησο του Σινά και πολλές άλλες πράξεις τρομοκρατίας ε, στην Αίγυπτο. Έχουμε επιθέσεις στους ε, κόπτες, χριστιανούς. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα φαινόμενα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουν δικαιολογία οι Αιγυπτιακές αρχές να διατηρούν θανατική ποινή. Ανησυχώ με μαζικές δίκες που γίνονται από τα Αιγυπτιακά δικαστήρια και πολλές θανατικές καταδίκες. Καλό τις Αιγυπτιακές αρχές να θέσουν τέρμα σε αυτές τις πρακτικές ε, και να ανακαλέσουν τις θανατικές ποινές. Επίσης θα πρέπει άμεσα να υπάρξει μορατόριο των εκτελέσεων. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατάρτιση θανατικής ποινής. Εμείς, Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδικάζουμε περίφραστα τις θανατικές ποινές. Πρέπει να τηρήσουν ε, η Αιγύπτιοι τις διεθνείς δεσμεύσεις τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Δεύτερο, Δεύτερος ε, ο κύριος Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, καθώ η Αίγυπτο ε, κάνει τη μετάβασή τη προ τη δημοκρατία, έχει πολύ, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρέ απειλέ εσωτερική ασφάλεια, όπω δείχνουν οι καταστρεπτικές επιθέσεις στο ίσως ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα στο Σινά και κατά των κοπτών, όπως είδαμε και στις χώρες μας, το να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της ασφάλειας και της τήρηση των ελευθεριών είναι πάντα δύσκολη. Ωστόσο, δικαίως εμείς θίγουμε τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό διεθνή εταίρο. Διαρκή η χρήση του στρατιωτικού η χρήση βασανιστήριων και η αυξανόμενη ε, χρήση της θανατικής ποινής είναι όλα αίτια για ανησυχία. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κλίση για περαιτέρω έρευνα στον, ε, για το θάνατο του Ιταλού υπήκου Τζούλιαν ε, Ρετζίνη που κατοικούσε στη Βρετανία και ένα μεγαλύτερη υπευθυνότητα από πλευρά των Αιγυπτιακών αρχών. Κυρία Σαργεντίνη, θέλει να Σα ερώτηση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε για αυτή τη μετάβαση προς τη δημοκρατία. Ε, εγώ δεν πιστεύω πως μπορούμε έτσι να εκτιμήσουμε την κατάσταση της χώρας. Είναι μια χώρα όπου υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος με πραξικόπημα πήρε την εξουσία και τους τελευταίους μήνες δολοφόνησε, σκότωσε 20, πάνω από 20 ανθρώπους. Για μας η θανατική ποινή είναι φρικτή και πάντοτε είμαστε αντίθετοι. Ζητάμε από τις χώρες πάντα να μην σκοτώνουν, να μην δολοφονούν τους ανθρώπους. Ε, και αυτό ακριβώς πριν τις εκλογές στην Αίγυπτο Ε, στις εκλογές ή θα ψηφίσουν για το ΣΥΣΥ Η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη δεν έχει καταδικάσει ακόμα τις δολοφονίες ε, της κυβέρνησης Σίση. ΣΥΣΥ. η Ευρωπαϊκή κυβερνησης ΣΥΣΥ. ειναι πλεον καιρος η ευρωπαικη επιτροπη να πάρει θέση απέναντι στα όσα γίνονται στην Αίγυπτο. Σάκε, ένα Α, όχι, με συγχωρείτε, ο κύριος Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα ε, συζητάμε και μια χώρα που έχει ξεπεράσει κάθε όριο στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για κράτος δικαίου. Από τότε που ο Σίση έχει την εξουσία, η Αιγυπτιακή εξουσία όχι μόνο έχει αυξήσει τις ε, καταδίκες σε θάνατο, αλλά έχει και αρχίσει και να τις εκτελεί. Σαν να μην αρκούσε αυτό, τους τελευταίους μήνες το φαινόμενο αυτό αυξάνεται με ε, αστρονομικούς ρυθμούς. Μια όξυνση της πλήρης κατάρρευση των αξιών του κράτους δικαίου ε, ε, παρακολουθούμε στην Αίγυπτο. Γι' αυτό σε αυτό το πλαίσιο ο συμπατριώτης μου Τζούλιο Ρετζένι ε, απήχθη και τελικά ε, δολοφονήθηκε. Δεν μπορούμε να το βρούμε ούτε και νεκρό, γιατί είναι εξαιρετικά ισχυρά τα οικονομικά συμφέροντα ε, συνεργασίας με την Αίγυπτο. Εάν οι Αιγυπτικές αρχές επέτρεψαν, επέτρεπαν να γίνει κάτι τέτοιο σε έναν ερευνητή που θα που θα τον έψαχνε η Δύση, δεν θέλω ούτε να φανταστώ ότι ο, τι επιφυλάσσει η τύχη η μοίρα στου Αιγύπτου υπηκό, οι οποίοι είναι τελείω άοπλοι και εγκαταλελειμμένοι στις ε, βουλές ενός ε, τυράννου. Δεν φτάνουν όμως αυτές οι ε, συζητήσεις, γιατί είπατε εκπρόσωποι φαίνεται να έχει παραιτηθεί σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Εμείς ως εγγυητές του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να μετατρέψουμε τα λόγια σε πράξεις. Τώρα η κυρία Σχάκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε συνάδελφοι, η καταστολή, η καταπίεση στην Αίγυπτο υπό τον στατηγό ΣΥΣ έχει δημιουργήσει μια ορολογιακή βόμβα. Κανεί δεν έμαθε τίποτα από την ιστορία. Εκτό που πνίγει τον ελεύθερο λόγο και περιορίζει τις ΜΚΟ, ε, εντυπωσιακό αριθμό εκτελέσεων. Πάνω από 2.000 έχουν εκτελεστεί από το 2014 και ε, ε, και 18 από την 1η του 2018 εκτός από αυτά βασανιστήρια, καταναγκαστικές καταθέσεις και κακομεταχείριση. Η Αίγυπτος έχει να αντιμετωπίσει θέματα ασφάλειας από την τρομοκρατία, αλλά η απάντηση ποτέ δεν είναι η κρατική η τρομοκρατία. Είναι πλέον καιρό, είπατε εκπρόσωπος, καθώς και τα ηγέτες των κατών μελών να τα πούν και να καταδικάσουν αυτές τις καταχρήσεις. Η σιωπή αυτή είναι κοφαντική. Είναι ενδιαφέρον να μιλάμε για έναν εταίρο, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Αν αυτό, αυτή η σχέση δεν βασίζεται σε κάποιες μήνυμα αξίες ε, που μας είναι κοινέ, τότε θα πρέπει να ε, διερωτηθούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Πόστο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε τις εκτελέσεις που γίνονται στην Αίγυπτο. Η θανατική ποινή αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή. Είναι η ίστατη, βίαιη, απάνθρωπη και υποβαθμιστική μεταχείριση απέναντι σε έναν, σε ανθρώπινο Καμιά πρόκληση, καμιά περίσταση Καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να αιτιολογήσει τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Η θέση του Ευρωκοινοβουλίου είναι η σε κατάργηση και αυτό υποστηρίζουμε. Ο διπλασιασμός των εκτελέσεων στην Αίγυπτο δεν είναι εξαίρεση όλα τα αυταρχικά ε, καθεστώτα χρησιμοποιούν ε, σε δυτικά δικαστήρια και συγκεκριμένες νόμους για να στοχεύσουν τις δραστηριότητε των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί μάλιστα δεν μπορούν να έχουν καν πρόσβαση σε ε, βοήθεια δικηγόρου ή έχουν ε, μπει στην απομόνωση και τους έχουν στερηθεί τα πιο βασικά τους προνόμια. Εγώ θα ήθελα να καλέσουμε τον ε, πρόεδρο Σίση να, καταργήσει, να σταματήσει τις εκτελέσεις και να καταργήσει τη θανατική ποινή. Στην κυρία Μογκερίνη λέω, πρέπει να υπερασπιστείτε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταδικάσετε τις εκτελέσεις. Τελευταία συντάκτρια είναι η κυρία Βερζιά. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλες οι ΜΚΟ μας ενημερώνουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ποτέ δεν είχαν τόσο καταπατηθεί στην Ένωση. 600.000 συλλήψεις, ε, ακόμα και 150 παιδιά τα τρία τελευταία χρόνια έχουν περάσει από στρατιωτικά δικαστήρια ε, και τα βασανιστήρια είναι καθημερινά. Οι υπερασπιστές δικαιωμάτων, ε, ΛΟΑΔΜΑ, δημοσιογράφοι είναι τα κύρια θύματα. Η προσφυγή στη θανατική ποινή δεν έχει πια όρια από ό,τι φαίνεται. Τρομοκρατία, κατοικία ασφάλεια, ε, εμπόριο ναρκωτικών, ε, δολοφονίες κτλ. Ο κατάλογος είναι μακρύς και είναι μια πραγματική δημιουργία. Πώς μπορεί να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Ε, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο όνομα μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης που δεν είναι και αυτά απόδεικτη. Ε, ωραία, τώρα οι ομάδες, ο κύριο Κέλλη από το ΕΛΚ. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ ισορροπημένο ψήφισμα το οποίο αναγνωρίζει τις δυσκολίες ε, που έχει ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις ε, που βιώσαμε προσφάτως, επιθέσεις κατά των κόπτικο της κοπτικής ορθόδοξης Εκκλησίας του Καθεδρικού Ναού και άλλες. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν είναι κατανοητό να αντιδρούν υπερβολικά οι αρχές, αλλά από την άλλη είναι απαράδεκτο όταν υπάρχουν ε, μαζικές ε, ε, δίκες, εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν με θανατική ποινή, ανθρώπους που βρίσκονται στη φυλακή μέχρι να φτάσει η στιγμή της δίκης τους για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και προβλήματα για τα πολιτικά και ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν οι Αιγύπτιοι να εξετάσουν το θέμα, να υπάρχει ένα μοραπτόριο για τη θανατική ποινή μέχρι την τελική κατάργησή της και ταυτόχρονα ε, να συνεχίσουν τη μάχη κατά της τρομοκρατίας οι Αιγύπτιοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Παντζέρη εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης 2017-2020 με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίγυπτος είχε δεσμευθεί να προωθήσει τη δημοκρατία, τις αμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει και του συντάγματός της και των διεθνών κανόνων. Αυτή η δέσμευση βεβαίως δεν τηρήθηκε και αυτό καταδεικνύουν οι ε, πολυάριθμες ε, θανατικές καταδίκες ε, που, τους τελευταίους μήνες που οδήγησαν στο θάνατο πολιτών που πριν είχαν υποστεί βασανισμούς και Χωρί ε, χωρίς καμία κοινοποίηση και ψευδοδίκε ενώπιον στρατοδικείων. Ε, αυτό το ε, τραγικό ε, γεγονός ε, συνέβη επανειλημμένος ε, κατά την κυβέρνηση του ΣΥΣΥ και είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια σταθερή εταιρική σχέση με τη χώρα αυτή με όλα όσα συμβαίνουν. Εκτός και αν ε, για λόγους realpolitik δεν ασχοληθούμε καθόλου με τα ανθρώπινα δικαιώματα και επομένω είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι ηθικά για όλες αυτές τις βαναυσότητες. Σίγουρα χρειάζεται σαφής δέσμευση για να μπορέσει να αλλάξει η Αίγυπτος από πλευράς Προέδρου του. Αλλιώς δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο αυτής εταιρική σχέση. Δράτω με δε τι ευκαιρίε να υπενθυμίσω ε, και τη συμπεριφορά ε, του καθεστώτο που είναι εκδικητική. Ε, Εμεί περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τον Ιταλό πολύ που δολοφονήθηκε πριν από δύο χρόνια στο Κάιρο. Και με αυτό το γεγονό καταδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια από πλευρά Αιγυπτιακών αρχών. Εξ ονόματο συστηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριο Βίστησεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να σας πω ότι δεν είδαμε να υπάρχει καμία εξέλιξη μετά την Αραβική Άνοιξη για την Αίγυπτο. Η μουσουλμανική αδελφότητα είναι ένας παράγων ο οποίος προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, το Αιγυπτιακό καθεστώς έχει προβλήματα, αλλά υπερβάλλει. Και πιστεύω ότι εδώ, όταν διαπιστώνουμε τι συνέβη στο Ιράν με τις διαδηλώσεις, όταν βλέπουμε επίσης και αντιδράσεις άλλων καθεστώτων και όταν έχουμε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Ε, εγώ σπαταλώ ενέργεια, μιλώ για την Κίνα, για το Ιράν, αλλά ε, για την περίπτωση της Αιγύπτου δεν μιλάμε κάθε τρεις μήνες. Θα πρέπει λοιπόν ε, να πούμε ότι η Αίγυπτος πρέπει να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τη δημοκρατία, αλλά να μην υπερβάλλουμε κιόλα. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από το πραξικόπημα του 13, το Μάρτιο, ε, θα γίνουν στην Αίγυπτο ε, ε, προεδρικές εκλογές που κατά ότι δεν θα έχουν αντιπολίτευση γιατί έχουν αποσυρθεί λόγω εκφοβισμού και συλλήψεων όλοι οι άλλοι υποψήφοι. Υποτίθεται ότι καταπολεμάται η τρομοκρατία και στο όνομα αυτής της προσπάθειας καταπνίγεται η κοινωνία των πολιτών, το δημοσιογραφικό κίνημα, το εργατικό κίνημα που παρόλα αυτά συνεχίζει να οργανώνει συλλαλτήρια και απεργίες. Πρόκειται για μια χώρα όπου τον τελευταίο μήνα εκτελέστηκαν 23 άτομα μετά από δίκη σε στρατοδικείο, χωρίς καμία εγγύηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά αποφασίζει να στρέψει αλλού το βλέμμα και να, να ε, ξεκινήσει τις επαφές της ε, παρά τις ε, κατάφρασης παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν απαιτούμε να αποφανθεί για αυτές τις παραβιάσεις, να απαγορεύσει τις εισαγωγές όπλων στην Αίγυπτο η Ένωση και να πάψει να νομιμοποιεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα εφόσον δεν γίνονται σεβαστά τα δημοκρατικά δικαιώματα τα πλέον θεμελιώδη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάρμπαρα Λοχμπίλερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Αίγυπτο καταδικάστηκαν σε θάνατο 2.000 άτομα και 81 έχουν ήδη εκτελεστεί. Και υπάρχουν φόβοι να αυξηθεί μαζικά ο ρυθμός των εκτελέσεων. Επίσης, η κατάσταση των δικαιωμάτων ε, στην Αίγυπτο είναι δραματική. Όσοι ασκούν επικρίσεις συλλαμβάνονται. Ε, δημοσιογράφοι, υπέρμαχοι δικαιωμάτων, αυθαίρετες κρατήσεις, ε, αγνοούνται άνθρωποι. Υπάρχουν έρευνε που λένε ότι υπάρχουν συστηματικά βασανιστήρια των κρατουμένων. Όλα αυτά είναι επονίδιστα. Πολύ επιφυλακτικά παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον 2017 υποτίθεται ότι αποφάσισε στο πλαίσιο του διαλόγου και της συμφωνίας σύνδεσης εκτός τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά παρόλα αυτά παρατηρούμε επιδείνωση κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει επομένως να κρυφτεί στα ωραία λόγια αυτά, ε, πίσω από τα ωραία λόγια της Αιγύπτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ασκήσει πίεση στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Καστάλδο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στις 26 Δεκεμβρίου 15 άνδρες που κατηγορούνταν για τρομοκρατία οδηγήστηκαν ε, ε, στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις Αιγυπτιακές Αρχές. Ε, εκείνη την ημέρα έσπασε ένα νέο ρεκόρ, τις περισσότερες εκτελέσεις σε μία ημέρα από το 1993. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάνω τους σημάδια από κάψιμο, από μαστίγωμα, ένδειξη βασανισμών, βάναυσων που και απαράδεκτων, εξαφανίσεις δημοσιά γράφων, αντιφρονούντων και διανοουμένων, όπως έγινε και με τον Τζούλιο Ρετζέρι, ο οποίος ε, σκοτώθηκε και υπάρχει μια ε, παγερή σιωπή για το τι του συνέβη. Και δεν υπάρχει και καμία εδώ ενώπιον αθώων παιδιών. Ε, δύο παιδιά 13 και 15 ετών απήχθησαν από το σπίτι τους και βρέθηκαν νεκρά μετά από μερικές μέρες στο χωριό τους. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται είναι και ευρωπαϊκά όπλα. Το εμπόριο και η Real Politik δικαιολογούν αυτή την ένοχη σιωπή των χωρών μα. Αυτή είναι η διαδικασία τη ασφάλεια και σταθερότητα που θέλουμε με την Αίγυπτο. Εγώ λέω όχι, θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μα να ζητήσουμε εμπάργκο όπλων και να ζητήσουμε αλήθεια και δικαιοσύνη για τον Τζούλιο Ρετζένη και για όλα τα αθώα θύματα αυτού του ε, βάναυσου καθεστώτος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βάιντεν Χόλτσερ έχει τώρα το λόγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια συζήτηση για την κατάσταση στην γειτόνα χώρα, την Αίγυπτο δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε τις πιέσεις βλέποντας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πραγματικά είναι απατηλό και επικίνδυνο να θεωρήσουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί στα ασφάλεια ε, μέσω της ε, τρομοκρατίας και της καταπίεσης. Ε, αυτό είναι επικίνδυνο και σίγουρα ό,τι γίνεται εκεί επηρεάζει και εμάς την Ευρώπη. Το κράτος δικαίου, δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο καλύτερος εγγύτης σταθερότητας και ασφάλειας. Γι' αυτό με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία βλέπουμε αυτή την αιμονή της Αιγύπτου με την θανατική καταδίκη την καταπολέμηση ε, της αρχής του συναθρίζεστε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε και με ευκαιρία τις επόμενες πρωτικές εκλογές ε, το θάρρος να ζητήσουμε ασκώντας πίεση περισσότερη δημοκρατία στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μπόιλαν. Ένα λεπτό. Ξανασυζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο. Καταδικάζουμε σήμερα όχι μόνο ε, τη θανατική ποινή, αλλά και την κλιμάκωση ε, της κατάστασης επί Προέδρου Πολλά είναι τα προβλήματα. Ο Ιμπραχήμ ο Ιρλανδός, μπορεί να πει από 26 Δεκεμβρίου έως 13 Ιανουαρίου να εκτελούνται πάνω από 10 άτομα, ε, τα Πολλοί είχαν ε, ε, καταδικαστεί από στρατοδικείο και οι δικηγόροι των εκτελεστάντων ούτε καν είχαν ενημερωθεί. Ε, ούτε οι οικογένειες των κρεμασμένων δεν μπόρεσαν να τους αποχαιρετήσουν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν το πτώμα, το σωρό του συγγενούς τους και δεν ξέρουν πού θα το βρουν. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η Αίγυπτος έχει υποχρεώσεις διεθνεί απέναντι ε, λόγω της Ένωσης, λόγω της Συμφωνίας σύνδεση δεν μπορεί να καταπατά και να καταπνίγει όλα τα δικαιώματα. Δεν ε, ε, πρέπει να σταματήσουμε εμείς να υποστηρίζουμε τους Αιγυπτίους γιατί αυτοί δεν έχουν φωνή για να το πράξουν. Ευχαριστώ. Η κυρία τώρα Νίνα Γκίλα. Όταν την τελευταία φορά τον Οκτώβριο συζητήσαμε την Αίγυπτο, η Κομισιόν περιέγραψε τις ε, προσδοκίες του Αιγυπτιακού λαού για ασφάλεια και οικονομική ευημερία. Εγώ έχω πραγματικές επιφυλάξεις για τη φύση της εταιρικής μας σχέσης τότε και τώρα ακόμη περισσότερο. Μιλάμε για πολύ μεγάλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ε, σχεδόν 40 εκτελέσεις το μήνα, 24 καταδίκες σε θάνατο, από στρατιωτικά δικαστήρια. Ε, ε, πραγματικά μπορείτε να μας περιγράψετε τον αντίκτυπο ε, που θα έχουν οι Αιγυπτικές αρχές αν δεν επιβάλλουν μορατόριο άμεσα για τη χρήση θανατικής ποινής και αν δεν αναθεωρήσουν τις νομοθεσίες τους για δίκαιες δίκες. Πότε θα πάψουμε να πουλάμε εξοπλισμούς ε, στο Αίγυπτο ώστε να σταματήσουν να βασανίζουν τον λαό τους και πότε θα γίνουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Ακόμα και αν δεν ε, θα, πρέπει να, γίνει, ε, δεν υπάρξει πλήρης κατάργηση της ανατικής ποινής, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές μας. Ο κύριος Φαρία.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 σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, χιλιάδες ε, διαμαρτυρώμενοι στην ε, συμβολική πλατεία τα Χρήρ ε, στο Κάιρο απέδειξαν τι συμβαίνει στην Αίγυπτο. Όμως θα γίνουν εκλογές σε λίγο και διώκονται ακτιβιστές, ΛΟΑΔΜΑ, υπερασπιστές των ανθρωπίνων ε, υπάρχουν μαρτυρίες για ε, βασανιστήρια και ε, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι θανατικές ποινές και οι εκτελέσεις. Έχουμε, έχουν τριπλασιαστεί οι θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν μέσα στο 2017 και μέσα στον Ιανουάριο 22 θανατικές ποινές εκτελέστηκαν αφού επιβλήθηκαν από στρατιωτικά δικαστήρια. Είμαστε η πρώτος οικονομικός εταίρος της Αιγύπτου και θα πρέπει να την υποχρεώσουμε να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα με άμεση πάυση της χρήσης της θανατικής ποινής. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Η κυρία Ιζαμπέλ Ντελμόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα θα εγκρίνουμε ένα κοινό ψήφισμα με σαφέ περιεχόμενο. Στην τρίτη χιλιετία, σε κανένα κράτο του κόσμου δεν μπορούν ακόμα να γίνονται βασανιστήρια, ε, συνοπτικέ εκτελέσει και παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτο οικονομικό εταίρο τη Αιγύπτου, αλλά δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια απέναντι σε βίαιη μεταχείριση. Μιλάμε για τον Τζούλιο Ρετζένι, ένα νεαρό ερευνητή που βάρβαρα βασανίστηκε και έπειτα δολοφονήθηκε στην Αιγύπτο. Ήταν παιδί αυτή τη Ευρώπη που βασίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που καταπατήθηκαν. Ίσως κάποιοι να ήλπιζαν ότι μετά από κάποιο χρόνο όλα αυτά θα είχαν ξεχαστεί. Αλλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σκοπεύουμε να σοπάσουμε και πάντα θα ζητάμε και μάλιστα έντονα για αυτή την ανθρωποκτονία να ε, διαλευκανθεί. Οι αρχές της Αιγύπτου θα έπρεπε μετά από δύο χρόνια να μας έχουν δώσει σαφή απάντηση που θα δώσουμε στην οικογένειά του στους φίλους του Τζούλιο αλλά και στα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά ότι είναι ασφαλής προορισμός η Αίγυπτος και καλός εταίρος. Πρόεδρος Πολτσακ. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. I já se připojuji ke svým kolegům, eh, pokud... Πρόεδρε, ε, σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να υποστηρίξω του συναδέλφους ε, ε, που μιλούν κατά της θανατική ποινή και μιλούν για συγκεκριμένες υποθέσεις. Πιστεύω πως υπάρχουν διπλωματικά εργαλεία για να πιέσουμε όχι μόνο τις, τις Αιγυπτικές Αρχές αλλά και την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη προσέγγιση προς τη θανατική ποινή. Δυστυχώ δεν έχουμε πολλούς εταίρους παγκοσμίω που να μπορούν να πιέσουν το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ε, τον ε, πρωτοπόρο ρόλο σε αυτή την υπόθεση και υποαίρεση να συνεχίσει τη συνεργασία με αυτή τη χώρα ε, το συζητάμε θα πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις χώρες που ε, δείχνουν ότι είναι πρόθυμες να συνεργαστούν όταν μιλάμε για την θανατική πίνη. Ε, διαφορετικά δεν θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί την κατάσταση, παρακολουθεί την κατάσταση στην Αίγυπτο στενά. Η άποψή μας για τη θανητική ποινή είναι ευρέως γνωστή. Η Αίγυπτος επιβάλλει θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι για μας αυτό αντιπροσωπεύει απαράδεκτη άρνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ακαιρεότητας. Στην Υποεπιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Αιγύπτου για τα πολιτικά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που έγινε στο Κάιρο τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ανησυχία της ε, στις Αιγυπτιακές Αρχές για την πρόσφατη εκτέλεση πάνω από 20 ατόμων και επαναλάβαμε την βασική μας θέση κατά της θανατικής πυλής. Ε, έγινε έκκληση προς την Αίγυπτο να περιορίσει τη ε, θανατική καταδίκη ε, το όπου είναι δυνατόν και να υπάρχει ένα μορατόριο με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής. Επιπλέον, ε, θα ρίνουμε την Αίγυπτο να λάβει συγκεκριμένα βήματα για να μην υπάρχουν στρατοδικεία για πολίτες και επίσης ε, να ε, ξαναδικαστούν οι πολίτες οι οποίοι δικάστηκαν από στρατοδικεία σε απλά δικαστήρια βάσει διεθνούς δικαίου για να υπάρχει δίκαιη δίκη. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέρω και μια σειρά από άλλα θέματα για ιστοσελίδες και οργανώσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σαφείς ανησυχίες όσον αφορά ε, το γεγονός ότι μπλοκάρονται ιστοσελίδες και υπάρχει πίεση προς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην θέση της για το Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου τον ε, Ιούλιο στις 17 του μηνός. Η θέση αυτή εκφράστηκε και στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Δήλωση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο σημείο 4, καθώς επίσης και στην ε, τελευταία υποεπιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου για πολιτικά θέματα που έγινε στο Κάιρο τον Ιανουάριο τον προηγούμενο μήνα. Επομένως, η, Αιγυπτο, η Αίγυπτος σίγουρα είναι βασικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, σημαντικός περιφερειακός παράγων η σταθερότητα και η ασφάλεια της χώρας είναι ζωτική σημασία όχι μόνο για τους ίδιους τους Αιγεπτίους αλλά και την ευρύτερη περιοχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μας. Είναι απόλυτη πεποίθησή μας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης ελευθερίας είναι πάρα πολύ σημαντικά για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος. Εκτιμούμε τις ε, δυσκολίες ε, και στεκόμαστε στο πλάι της Αιγύπτου ε, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό βασίζεται σε καθολικές αξίες και τα συζητάμε τακτικά με τους Αιγυπτίους εταίρους μας στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλία για τις προτεραιότητες ε, της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, Αιγύπτου που όπως γνωρίζετε ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2017. Επικεντρωνόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και αυτές είναι οι αρχές που διέπουν τη δράση μας στο εξωτερικό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προωθούμε ενεργά και να προασπιζόμαστε αυτές τις αρχές ενεργά στις επαφές μας με την Αίγυπτο, όπως κάνουμε και με όλους τους εταίρους μας ε, ανά τον κόσμο. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι δύσκολη, αλλά προσπαθούμε πολύ προκειμένου να πιέσουμε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Πέντε προτάσεις ψηφίσματος υπάρχουν για την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης.